Colleagues, καθίστε παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς ορίζω όλους τους βουλευτές και τους καλεσμένους μας σε αυτή την ολοήμερη συνεδρίαση της ΕΝΤΕ. Έχουμε τα πρώτα σημεία μαζί με την ΑΦΕΤ και τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες. Θα ήθελα ως συνήθως να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο, ως συνήθως. Και ως προς τη διερμηνία έχουμε δώσει προτεραιότητα ε, στις γλώσσες των τακτικών μελών Θα ήθελα να υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, άρα υιοθετείται η μερίσια διάταξη. Και τώρα θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι σήμερα θα υιοθετήσουμε και τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου, της 3ης Δεκεμβρίου του 2018. Η προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων είναι μέχρι σήμερα, το τέλος της συνεδρίασης. Αν έχετε σχόλια, να τα υποβάλλετε στη γραμματεία. Μια μικρή ανακοίνωση επίσης. Ευχαριστώ τους συντονιστές και τους βοηθούς μου, τους αναπληρωτές μου που βοήθησαν και εμένα και τη, γραμμα... και τη γραμματεία επίσης ευχαριστώ ε, που με βοήθησαν και με στήριξαν κατά την μακρά απουσία μου γιατί έπρεπε να εγχειριστώ. Ήταν απαραίτητο αυτό. Σας ευχαριστώ πραγματικά για τη βοήθειά σας. Όλους όσους ε, με αντικατέστησαν ε, στην Προεδρία, το, την κυρία Μούντι, τον κύριο Στετίνα και τον κύριο Γκάλερ που είναι ο συντονιστής του ΕΛΚΑ. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι με αντικατέστησαν και προέδρευσαν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ΕΝΤΕ. Θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως και ολόκληρη τη γραμματεία για τη βοήθεια που μου έδωσε, το προσωπικό βεβαίως, οι, τους συμβούλους και τους δικούς μου βοηθούς. Ήταν δύσκολη η περίοδος, αλλά τώρα είμαι καλά πάλι, όπως βλέπετε. Και χωρίς να καθυστερήσω περαιτέρω, θα ήθελα να δώσω το μικρόφωνο στην κυρία Τεμπράφκα Σουίτ, αντιπρόεδρο της ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ, Άννα. Καλημέρα σε όλους. Είναι μια κοινή συνεδρίαση σε ΑΦΕΤ. Το τέταρτο σημείο στην ημίσια διάταξη είναι τα συμφέροντα ασφαλεία τη Κίνα και η επιρροή τη στην Αφρική. Θα κάνουμε μία ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Χωακίν Τάσο Βιλαλόγκα, που είναι ο αναπληρωτή τμήματάρχη Παναφρικανικών Υποθέσεων τη ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και τη κυρία Βαλερίνη Κε, επικεφαλή προγράμματο Ασία του Ιδρύματο Στρατηγική Έρευνα. Θα ήθελα να παρουσιάσω αυτό το θέμα. Η Κίνα έχει τεράστια επιρροή στην Αφρικανική Ήπειρο τα τελευταία 15 χρόνια με μεγάλες επενδύσεις, δάνεια σε υποδομές και φυσικούς πόρους σε αφρικανικές χώρες ε, που συχνά δεν έχουν πρόσβαση στην ε, χρηματοδότηση. Αυτό γίνεται χωρίς όρους και χωρίς να συνδεθούν οι επενδύσεις αυτές με αξίες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες. Οι υποδομές της Αφρικής ε, δεν είναι σε καλή κατάσταση, έχει τεράστιες ανάγκες και είναι πολύ ελκυστικό για τις χώρες της Αφρικής ε, να δέχονται ε, χρηματοδότηση χωρίς όρους. Οι ποσαχάριες χώρες έχουν ανάγκες ε, κάθε χρόνο 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα υποδομών και να φτάσουν σε ηλεκτροδότηση 100% και 100% πρόσβαση σε πόσιμο νερό και αποχέτευση. Η χρηματοδότηση των από την Κίνα μπορεί να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμα κέρδη και δημοτικότητα αυτών των κυβερνήσεων. Αλλά αυτό έχει κινδύνους, διότι αυτές οι χώρες μπορεί να πέσουν σε μακροπρόθεσμη χρέωση και εξάρτηση από τους δανειστές στην Κίνα. Αυτό έχει συμβεί με τους γείτονες της Κίνας στην Νοτιοανατολική Ασία, παρότι οι χώρες αυτές έχουν μεσαίο εισόδημα και έχουν παρόλα αυτά τεράστια χρέωση και άνοιγμα απέναντι στην Κίνα. Ταυτόχρονα, η κινέζικη παρουσία έχει προωθήσει το εμπόριο κινέζικων προϊόντων στην Αφρική. Υπάρχει ανησυχία ότι η εισρωή κινέζικων προϊόντων και πάνω από 10.000 κινέζικων ε, εταιριών στην Αφρική έχουν περιορίσει το χώρο για τους ντόπιου επιχειρηματίες. Εμείς ως Ευρωπαίοι θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση των χωρών της Αφρικής για τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα και κινδύνους αυτής της πολιτικής δανεισμού και να ενθαρρύνουμε την, τις επενδύσεις της Κίνας να βοηθήσουν την ανάπτυξη της Αφρικής και την βιομηχανία της, ε, ούτως ώστε να ανέβει στην αξιακή αλυσία αλυσίδα η Αφρική, στην αλυσίδα δηλαδή προσθέμενης αξίας ε, και να μην είναι απλώς μια πηγή πρώτων υλών. Η Κίνα έχει δώσει 85 δισεκατομμύρια δολάρια στην Αφρική ανάμεσα στο 2013 και στο 2017 και έχει δεσμευτεί να δώσει άλλα 60 δισεκατομμύρια σε δάνεια επιχορηγήσει επενδύσει στην Αυστρία τα επόμενα χρόνια. Η Αφρική γίνεται όλο και πιο νευρική για αυτό το χρέο που έχει απέναντι στην Κίνα και το Φόρουμ Συνεργασία Κίνα-Αφρική ε, πέρυσι το φθινόπωρο δεσμεύτηκε να αυξήσει οι Κινέζοι μέσα από αυτό ε, δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τη βοήθεια και τις επενδύσεις στην Αφρική ε, και να δώσουν βοήθεια ε, για επενδύσεις, εμπόριο, για το περιβάλλον, για την υγεία και την ασφάλεια. Ήταν μια σύντομη εισαγωγή αυτή. Ο κύριος Χουακίν Τάσο Βιλαλόγκα, ο οποίος είναι απλωτής τμήματάρχης Παναφρικανικών Υποθέσεων, είναι εδώ. Λοιπόν, θα κάνουμε πρώτα μια παρουσίαση και μετά σχόλια. Εγώ διάβασα τις σημειώσει μου. Η κυρία Βαλερή λοιπόν θα κάνει την πρώτη παρουσίαση που είναι επικεφαλής του προγράμματος Ασίας του Ιδρύματος Στρατηγικής Έρευνας. Ε, εσείς πρώτοι. Θα ήθελα να κάνω μία προσθήκη. Λυπάμαι πάρα πολύ που επαναλαμβάνω και πάλι πως το θέμα είναι ε, τα συμφέροντα ασφάλειας της Κίνας και η επιρροή της Κίνας ε, στην Αφρική. Οπότε και πάλι ε, συζητάμε εδώ τις δραστηριότητες της Κίνας. Οπότε αυτό συνδέεται απόλυτα Ε, με τα θέματα της ανταπρεπίας ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και γι' αυτό θα καλωσορίσω τον κύριο Λάινεν που είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας αυτής και νομίζω ότι μετά τις παρουσιάσεις που θα ακούσουμε από τους συμμετέχοντες στο πάνελ θα μιλήσετε κι εσείς γιατί υπάρχει το θέμα αυτό, η, τα συμφέροντα και οι επιλές για την ασφάλεια από πλευράς Κίνας είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει σε πάρα πολλές ε, συναντήσεις της δικής μας επι υποεπιτροπής και έχουμε ε, εστιάσει κυρίως ε, στην κυβερνοασφάλεια και πώς αυτή σχετίζεται με τις κινέζικες δράσεις, όπως επίσης με την ελευθερία πλοήγησης και πιο συγκεκριμένα με τις κινέζικες δράσεις και δραστηριότητα στην ε, θάλασσα της Ανατολικής Κίνας. Επισκεφτήκαμε την Ιαπωνία και πέρσι και αυτό αποτέλεσε ένα μεγάλο κομμάτι των συζητήσεών μας. το έχουμε ξαναπεί συχνά και βέβαια οι δικοί μας συμμετέχοντες στο πάνελ αποφάσισαν να αντιστρέψουν τη σειρά των παρουσιάσεων, οπότε θα ζητήσουμε την κυρία Νικέ να λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Θα κάνω λοιπόν μια παρουσίαση στα γαλλικά και θα ξεκινήσω πιο σφαιρικά μιλώντας για τα αφρικανικά κινέζικα συμφέροντα και όχι μόνο από στρατιωτική πλευρά, αλλά ήθελα να σας δείξω πως αυτή τη στιγμή με την Κίνα και όχι μόνο με την Κίνα, αλλά συγκεκριμένα με το Πεκίνο, αντιμετωπίζουμε μια πολύπλευρη στρατηγική, η οποία κινητοποιεί μια σειρά εργαλείων, όπως αυτά τα οποία αναφέρατε, και που ε, αλληλοενισχύονται έτσι ώστε να προωθήσουν τα συμφέροντα του Πεκίνου στην Αφρικανική Ήπειρο. Και θα κλείσω την παρουσίασή μου ε, προσπαθώντας να κάνω και ε, μία αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κίνα στην Αφρική και εδώ θα συμπεριλάβω ε, και ίσως αυτό θα απηχηθεί από τις αφρικανικές χώρες οι οποίες ευιστοποιούνται για το θέμα της υπερβολικής εξάρτησης και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει αυτά από την Κίνα. Εδώ και 20 χρόνια, που είναι μια σύντομη περίοδος, η Κίνα είναι πια σήμερα ο πρώτος οικονομικός εταίρος της Αφρικανικής Υπήρου, αν συμπεριλάβουμε και την Βόρεια Αφρική, πρώτος επενδυτής 200 δις ε, ε, δολάρια για το 2017 τα δούμε σωρευτικά, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είναι ζωτική σημασία επενδυτή για τις περισσότερες αφρικανικές χώρες, κυρίως στην ενέργεια και την υποδομή. Στα θέματα αυτά θα επανέλθω. Η Κίνα επίσης είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Αφρικής και οι συναλλαγές με την Αφρική έχουν αυξηθεί ε, σημαντικά και έχουν όλο και περισσότερο βάρος και για την Κίνα την ίδια. Στην αρχή της ε, χιλιετίας οι συνοαφρικανικές εμπορικές συναλλαγές ήταν το 4% του συνόλου ε, των κινέζικων και το 2017 έχουν φτάσει το 13% των εξωτερικών εμπορικών συναλλαγών της Κίνας. Κατανοείται, λοιπόν πως δεν είναι αμεληταίο για την Κίνα και το στοιχείο αυτό και βέβαια για τους Κινέζους η αφρικανική αγορά γίνεται όλο και πιο σημαντική. Παρόλο που πάντα θα πρέπει να θυμόμαστε πως αυτή η αφρικανική αγορά είναι αγορά αναπτυσσόμενων χωρών και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις μεγάλες εμπορικές δυνάμεις και τις αγορές αυτών που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ. Και αυτό εξηγεί γιατί το Πεκίνο σήμερα ανησυχεί για τις εμπορικές τριβές που έχει με την Ουάσιγκτον σε διπλωματικό, ε, σε διπλωματικό επίπεδο, να σας πω παράλληλα, πως είχαμε μία αύξηση ε, των ε, συζητήσεων από τη δεκαετία του 90. Να σας πω πως Εκεί έγιναν οι πρώτες επισκέψεις Κινέζων αξιωμετούχων στην Αφρική για να προσπαθήσουν να αυξήσουν το, την παρουσία τους εκεί και ο πρόεδρος πήγε τον Ιούλιο του 2018, Ζιπίνγκ, ε, στην Αφρική, πήγε ε, Μαυρίκιο, πήγε Σενεγάλη και πήγε και στην ε, διάσκεψη των BRICS, που είναι η Ρωσία, η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία και η Νότιος Αφρική. Στην Ήπειρο αυτή λοιπόν έγινε λοιπόν τον Ιούλιο του 2018 η σχετική συνάντηση στην ε, Νότιο Αφρική και συμμετείχε και ο πρόεδρος της Κίνας. Να σας πω λοιπόν πώς Υπάρχουν και προσωπικές επαφές μεταξύ αφρικανικών χωρών και Κίνας με σχέσεις οικονομικές, με σχέσεις αρχηγών αφρικανικών κρατών οικονομικές με τη χώρα αυτή και συμμετοχή σε διάφορα φόρουμ συνεργασίας κινέζο-αφρικανικών ε, επαφών και πρέπει να σας πω πως αυτές οι συναντήσεις γίνονται μια φορά στην Κίνα και μια φορά σε κάποια αφρικανική χώρα. Θα επανέλθω αργότερα. Η στρατιωτική παρουσία των Κινέζων στην Αφρική αυξάνεται αυξάνεται είτε μέσω διμερών ε, ε, συμφωνιών είτε σε πολυμερές επίπεδο μέσω της Αφρικανικής Ένωσης και το 2015 η Κίνα για πρώτη φορά υπέγραψε ε, μια εταιρική σχέση για την ασφάλεια και την ειρήνη με την Αφρική. Είναι η πρώτη αυτού του είδους και δείχνει τη σημασία που έχει ακόμα και σε επίπεδο στρατιωτικό και επίπεδο ασφάλειας τη σημασία που έχει η Αφρική για την Κίνα. Επίσης, συμμετοχή μαζική της Κίνας στις αποστολές του ΟΗΕ για την διατήρηση της ειρήνης, ε, για τη μάχη ε, κατά της ε, πειρατείας στον κόλπο του Άντεν και το 2015 επίσης η Κίνα αποφάσισε μέσω αυτής της εταιρική σχέσης για την ασφάλεια και την ειρήνη που, στην οποία προανέφθηκα ο πρόεδρος Σιν Πινγκ άνοιξε ένα νέο σκέλος βοήθειας κινέζικης προς την Αφρική για να δημιουργηθεί μια αφρικανική ομάδα ταχείας κρούσης για να αντιμετωπίζει αφρικανικά στρατιωτικά σε εισαγωγικά προβλήματα. Αυτές λοιπόν οι, όλες, όλα αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται μεταξύ τους και αποδεικνύουν πως υπάρχει μια πραγματική αφρικανική στρατηγική την οποία εξαπλώνει και εξεδιπλώνει η Κίνα με στοιχεία μεταξύ τους συμπληρωματικά. Έχουμε κρατικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν, έχουμε ατομικέ επιχειρήσεις, έχουμε τον πολιτιστικό, το στρατιωτικό, τον οικονομικό κλάδο και, όλες αυτά, και όλα αυτά ε, είναι πολύ πετυχημένα γιατί γίνεται, ένας πολύ, ε, γίνεται μια πολύ δυναμική προώθηση ε, σε συλλογικό αλλά και σε μεμονωμένο επίπεδο με μικρές επιχειρήσεις για παράδειγμα και μην ξεχνάτε και το ότι η Κίνα χρησιμοποίησε το γεγονός ότι οι άλλες μεγάλες δυνάμεις μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου έδειξαν σε ένα βαθμό διαφορία για την Αφρική, οπότε πρέπει να το αναγνωρίσουμε η Κίνα μπήκε ε, να καλύψει ένα κενό ακόμα και σε επίπεδο βοήθειας με ε, κονδύλια για την επένδυση στην Αφρική. Και αυτό αποδεικνύει γιατί αυτή η διοίκηση της ε, Κίνας στην Αφρική ήταν τόσο πετυχημένη. Σε οικονομικό επίπεδο, όπως σας είπα, η στήριξη από πλευράς κοινωνιστικού κράτους είναι ιδιαίτερα υψηλή. Κινητοποίησε λοιπόν ε, κονδύλιο πολύ περισσότερο από άλλες μεγάλες δυνάμεις. Έχουμε πολλές κινέζικες επιχειρήσεις και βέβαια πολύ, πολύ οικονομικό ρεαλισμό χωρίς τις δικές μας αιρεσιμότητες στην Κίνα αναλαμβάνουν κινδύνους τώρα πρόσφατα με έναν τρόπο ε, πολύ πιο εύκολο σε εισαγωγικά από ότι αναλαμβάνουν τον κίνδυνο αυτό άλλες χώρες. Είναι, αυτό είναι, ε, συμπεριλαμβάνει και οικονομικούς κινδύνους και για την διακυβέρνηση σε εισαγωγικά ε, ε, Πρέπει να σας πω πως ε, εδώ γίνεται μια μάχη κατά τη διαφθοράς ε, στην Κίνα, αλλά αντιμετωπίζουμε διαφορετικό τρόπο τη σύναψη συμβάσεων με κάποιες ε, χώρες στην Αφρική και όχι μόνο, έτσι ώστε στο θέμα αυτό να έχουν ακόμα μεγαλύτερες ευκολίες. Από το 2015 και μετά η Αφρική αποτελεί κομμάτι της διαδρομής του μεταξιού και αυτής της στρατηγικής της Κίνας που ε, μέσω ενός ιδρύματος έχει σκοπό να κινητοποιήσει την Αφρική ε, και Εδώ επικρίθηκε το Πεκίνο γιατί όταν μιλήσαμε για την αξία της παραγωγής, για τις συνθήκες της παραγωγικής, ε, επειδή άκουσα ακριβώ αυτή τη επικρίση του Πεκίνο, αποφάσισε να βοηθήσει την εκβιομηχάνηση τη Αφρική με κάποια βιομηχανικά και ερευνητικά πάρκα, τα οποία, για παράδειγμα, στο Ντακάρ, στον Κικάλι, στη Ρουάντα, στήθηκαν σύμφωνα με τα αντίστοιχα κινέζικα στην Κίνα, έτσι ώστε να υπάρχει μετεγκατάσταση κινέζικων επιχειρήσεων, μια και ξέρουμε ποιο είναι το μισθολογικό κόστος αυτή τη στιγμή στην Κίνα και να γίνονται ε, εξαγωγές από τις πολύ φτωχές αφρικανικές χώρες προς τρίτες χώρες με έναν τρόπο που να τους ωφελεί οικονομικά. Άρα λοιπόν είδατε πως εδώ η Κίνα παρουσιάστηκε ε, στο να παρουσιάστηκε σαν να συνεισφέρει και το κάνει σε κάποιο βαθμό ε, στην εκβιομηχάνηση ε, των ε, φτωχών αφρικανικών χωρών. Δεν είναι μόνο όμως οικονομικές οι σχέσεις, είναι και ιδεολογικές. Γιατί αν ακούσετε τις δηλώσεις της Κίνας για την Αφρική θα μιλήσουν πάντα Ε, για τον διάσημο Κινέζο εξερευνητή που έφτασε στην Αφρική το 14ο αιώνα, για την παλαιότητα Κινέζικων και Αφρικών ε, ε, σχέσεων και επίσης για το γεγονός ότι και οι δύο χώρες έχουν αντιμετωπίσει την απεικιοκρατία. Και βλέπετε πως αυτό ε, αναφέρεται πάντα σε σχέση με το τι έκαναν οι παλαιότερες ε, μητροπόλεις των χωρών που είχαν απικείς ε, στην Αφρική και αυτό συγκρίνεται με την Κίνα. Να σας πω λοιπόν πως η στρατηγική της Κίνας αυτή τη στιγμή ε, δεν είναι καινούρια. Είναι μια στρατηγική που ξεκινά από το κύμα ανεξαρτησίας ε, των χωρών στην Αφρική που έχει στηριχθεί από την Κίνα και για το Πεκίνο αυτή η προϊστορία αποτελεί ένα πολιτικό κεφάλαιο για την σημερινή πολιτική ηγεσία και αυτή η ιστορική φιλία μεταξύ Αφρικής και Κίνας ε, που ιδρύει αυτές τις σχέσεις ε, ε, νότου με νότου, που είναι εποφελής και για τις δύο πλευρές, χρησιμοποιείται από αυτό το σε εισαγωγικό νεοεμπεριλιστικό, την νεοεμπεριλιστική πολιτική της Κίνας, για να έχει μεγαλύτερη επιρροή στην Κίνα. Θα θυμόσαστε τις περίφημες πέντε αρχές της ειρηνικής συμβίωσης. Αυτό είχε ε, ε, ε, εγκαθιδρυθεί την εποχή που είχαμε αυτή τις προσπάθειες απελευθέρωσης τη Αφρικής και πάντοτε κυριαρχούσε στις σχέσεις Κίνας με τις αφρικανικές χώρες. Και εκεί βασίζεται και σήμερα η κινέζικη βοήθεια προς τις αφρικανικές χώρες με πολλές δωρεές γιατί νομίζω ότι αυτή την τακτική θα ακολουθήσει και η μελλοντική πολιτική της Κίνας στη χρηματοδότηση της Αφρικής. Ιδεολογικά η επιτυχία του κινέζικου μοντέλου που μιλά για οικονομική ανάπτυξη με σταθερότητα έτσι το λέει το Πεκίνο, που βασίζεται σε μια αυταρχική πολιτική, έρχεται σε βασική αντίθεση με το δημοκρατικό ευρωπαϊκό μοντέλο που βασίζεται στις καθολικές παγκόσμιες αξίες και στο δημοκρατικό σύστημα όπως είναι στη Δύση, το οποίο στην Κίνα θεωρείται πως είναι λιγότερο αποτελεσματικό και πως δημιουργεί αναταραχές. Και αυτό το χρησιμοποιούν όταν κάνουν επαφές με τους αφρικανικούς εταίρους. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για εκδημοκρατισμό των διεθνών σχέσεων με τη δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας τάξης ε, με έναν τρόπο που συστηματικά προωθεί το Πεκίνο όπου μιλά για ιδεολογική κινητοποίηση, για εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος που είναι ε, πιο φιλικό για να γίνει μια μεγάλη και νομιμοποιημένη ε, δύναμη στο παγκόσμιο επίπεδο η Κίνα που θα υπηρετεί τα δικά της στρατηγικά συμφέροντα. Να σας πω πως ο πρόεδρος Σιπίνγκ πρόσφατα είπε η Κίνα παραπέμπω, ήταν και θα είναι ε, πάντα υπέρ των ε, χωρών αυτών και εναντίον όσων τους κτυπούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η δήλωση αυτή ενισχύεται από το project το δρόμο του μεταξιού που βασίζεται και σε ιδεολογικά και σε ε, οικονομικά, σε κοινωνικούς πυλώνες. Τώρα, για τα οικονομικά συμφέροντα, νομίζω ότι σας ανέφερα αρκετά προηγουμένως, να σας πω πως είναι και διαφοροποιημένα ε, αυτά τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά βασίζονται κυρίως το γεγονός πω υπάρχει οικονομική συμπληρωματικότητα. Η Κίνα χρειάζεται ακόμα πρώτε ύλε, χρειάζεται ενέργεια που προέρχεται από τι Αφρικανικέ χώρε, παρόλο που έχει ε, κάπως επιβραδυνθεί η, η κινέζικη ανάπτυξη. Το 2017 το 20% ε, του ε, πετρελαίου του ε, το εισήγαγε από την ε, Αφρική η Κίνα από την Αγκόλα και είναι ο τρίτος πάροχος πετρελαίου προς την, ε, Αφρική, προς την Κίνα μετά την Ρωσία και τη Σαουδική ε, Αραβία. Σας μίλησα για τα 200 δις και να σας πω πως το 80% βασίζεται στις συναλλαγές με πρώτες ύλε και με ενέργεια, ενεργειακά προϊόντα, τα υπόλοιπα έπονται. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, πολύ μιλήσαμε για την εταιρεία Huawei ε, και για το γεγονός πως είναι πάρα πολύ παρούσα στην Αφρική, δημιουργεί υποδομές για τις επικοινωνίες, είχαμε και τα πρόσφατα στον τύπο. Στην υψηλή τεχνολογία η Κίνα έχει αναπτύξει την παρουσία της στην Αφρικανική Ήπειρο και νομίζω ότι αυτό συνδυάζεται απόλυτα ε, και με τα σιδηροδρομικά project. Μου είπαν να τα πω πιο γρήγορα. Λοιπόν, τα στρατηγικά συμφέροντα δεν θα μιλήσω για την ε, Ταϊβάν, γιατί βέβαια είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά δεν είναι πια το πιο ουσιαστικό. Να σας πω πως η αφρικανική πολιτική της Κίνας της δίνει την ευκαιρία να ενισχύσει την δύναμή της στην παγκόσμια δικυβέρνηση. δηλαδή είναι αυτοί οι νέοι κανόνες που σύμφωνα με την Κίνα θα είναι πιο προσαρμοσμένοι στο να επιτρέψουν την ανάπτυξη χωρών όπως ε, αυτών που είναι στην Αφρικανική Ήπειρο. Το οικονομικό μοντέλο της Κίνας επίσης είναι ο τρόπος ανάπτυξης ε, ε, που νομιμοποιεί την ηγεσία στο να παραμείνει στην εξουσία και τέλος για να επανέλθω σε ένα θέμα το οποίο συνδέεται πιο στενά με το στρατιωτικό σκέλος και είναι και αυτό σημαντικό να σας πω πως στα πλαίσια μια πιο ε, ευρείας στρατηγικής για την Κίνα. Εδώ μιλάμε για την ε, άμυνα των οδών επικοινωνίας ε, μεταξύ Αφρικής και Κίνας, γιατί έχουν πετρέλαιο, έχουν πρώτες όλες, πρέπει να εξασφαλίσουν πως τα φτάνουν, με κάποια εξέλιξη την οποία όλοι είδαν το 2017 για πρώτη φορά, και αυτό αποτελεί ένα πολύ διαφορετικό ε, ε, στοιχείο για την Κίνα, άνοιξε στρατιωτική βάση στο Τζιμπούτι, ε, πρώτη φορά το έκανε, δίπλες σε άλλες δυνάμεις, για να υπερασπιστεί τα, κινη... τα κινέζικα συμφέροντα. Θα μπορούσα αργότερα να μιλήσω και για τις στρατιωτικές ειρηνευτικές ε, αποστολές, πολύ σημαντικό για το Πεκίνο, με τον τρόπο αυτό αναπτύσσουν ε, τις δυνατότητες που έχουν συνεργασία σε αφρικανικό έδαφος και να σας πω πως ένα σημαντικό στοιχείο είναι, και αυτό είναι ουσιαστικό, είναι ο δεύτερος πολιτής ε, όπλων στην Αφρική και αυτό συμπεριλαμβάνεται ελαφριά όπλα έχει υπογράψει τη σύμβαση ε, η Κίνα και βεβαίω αυτή η παροχή όπλων δημιουργεί πρόβλημα σε χώρες εύθραυτη όπου τα όπλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν από ένοπλες ομάδες ε, οι οποίες θα έχουν πρόσβαση σε αυτά. Τώρα, να κλείσω λέγοντας πως ο κίνδυνος ο οποίος δημιουργείται για την Κίνα είναι ο εξή. Έχει πολλά συμφέροντα, ενισχυμένα συμφέροντα, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι για το Πεκίνο. Δηλαδή, οι κατηγορίες της νεοαπικιοκρατίας. Κάτι το οποίο ακούγεται σε επίπεδο αφρικανικών πληθυσμών. Και υπάρχει και αυτό το ρήγμα μεταξύ των Αφρικανικών ελίτ και της κοινωνίας των πολιτών που δεν είναι πάντα τόσο έτοιμες ε, στην τόσο στενή συνεργασία με την Κίνα. Επίσης, η εκμετάλλευση των πρώτων υλών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο καταγγέλλεται συχνά ε, και είναι ένα θέμα συζητήσεις ε, μεταξύ Κίνας και Αφρικής. Και επίσης, γιατί είναι τόσο ελκυστική η Κίνα στην Αφρική, το γεγονός πως έχει ε, οικονομικό και οικονομική και εμπορική ισχύ, αλλά κάποιες χώρες ανησυχούν από τη μεγάλη εξάρτηση που έχουν από την κινέζικη αγορά, δηλαδή αγκόλα, πετρέλαιο και αυτό τις κάνει ακόμα πιο εύθραυστες, όπως συμβαίνει και με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και η επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κίνα αυτόματα σημαίνει και επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Αφρική. Για παράδειγμα, Είχαμε μία εχμή το 2014 215 ε, δις δισεκατομμύρια. Έχουν μειωθεί ε, σήμερα και αυτή τη στιγμή το 25% των καταναλωτικών τους αγαθών τα εισάγουν από την Κίνα αυτές οι χώρες και με τον τρόπο αυτό καταγγέλνουν το γεγονός πως καταστρέφονται οι ε, τοπικές επιχειρήσεις και βιομηχανία. Τέλος, για το Πεκίνο έχουμε ένα μεγάλο κίνδυνο πως είναι ο τεράστιο αριθμό Κινέζων υπηκών στην Αφρικανική Ήπειρο, δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία, αλλά μιλάμε για πάνω από ένα εκατομμύριο υπηκό ε, τουλάχιστον. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό να τον λαμβάνει υπόψη η Κίνα, γιατί έγιναν επιθέσεις κατά ε, κινέζικων περιουσιακών στοιχείων ε, και υπηκών στην Αφρική, κυρίως στο Μαλί. Θυμόσαστε τι έγινε στη Λιβύη και θέλει αυτή τη στιγμή... συγγνώμη κυρία μου, αλλά Μιλάτε πολύ γρήγορα. Ναι, αλλά έχω τόσα να πω. Θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά. Το τελευταίο, η Κίνα έχει την υποχρέωση, ή τουλάχιστον αισθάνεται την υποχρέωση σήμερα, να δικαιολογεί το γεγονός ότι ε, ε ξεδιπλώνει αυτή την στρατιωτική ισχύ στην Αφρική, ε, γιατί πρέπει να προστατεύσει άμεσα ε, περιουσιακά στοιχεία υπηκόους και να έχει τη δυνατότητα διάσωσης ε, παρόλο που αυτό ακόμα ε, σε πραγματικό επίπεδο δεν μπορεί να το καταφέρει. Για να το πω λοιπόν, ε, κλείνοντα, είναι ένα τοπίο ανισχυτικό, με, με πολλή εξάρτηση, με μια μεγάλη εξάπλωση τη κινέζικη παρουσία στην Αφρική, ακόμα και στρατιωτικά, που ανταποκρίνεται σε κάποιε προσδοκίε των αφρικανικών χωρών και μια πρόκληση για εμά. Μια άμεση πρόκληση για να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε αυτήν την κινέζικη παρουσία. Σα ευχαριστώ πολύ. Στι ερωτήσει, αν θέλετε, θα απαντήσω και στα αγγλικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χωακίν Τάσο Βιλαλόγκα, ε, αναπληρωτής τμήματάρχης τη ε, Παναφρικανική Παναφρικανικής στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος εγώ. Η ίδια η έννοια της αλληλεξάρτησης ε, αυξάνει τη στρατηγική σημασία της Αφρικής και τη βάζει πιο ψηλά στις προτεραιότητες μας. Ε, στο Αμπιτσάν το Νοέμβριο του 2017 είχαμε την πέμπτη διάσκεψη. Οι Αφρικανοί και Ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύτηκαν ε, για τέσσερις ε, στατικές προτεραιότητες. Επένδυση στους ανθρώπους, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση των νέων, ε, δεξιότητες και ανώτατη εκπαίδευση. Το δεύτερο, διακυβέρνηση ασφάλεια. Τρίτο, κινητικότητα και μετανάστευση. Και τέσσερα, κινητοποίηση επενδύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη και μετασχηματισμό της Αφρικής. Όπως γνωρίζετε, έχει μια φιλόδοξη ατζέντα περιφερειακής ολοκλήρωσης η Αφρική. Με μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών για όλη την Αφρικανική Ήπειρο, που όπως γνωρίζετε τώρα υπογράφεται και κυρώνεται από μεγάλο αριθμό αφρικανικών χωρών. Επίσης, κάνουν και μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε ε, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης να γίνουν πιο αποτελεσματικά, πιο λειτουργικά για να εξασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην Αφρική. Και με ένα ταμείο Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής, όπως γνωρίζετε, που χρηματοδοτεί ε, την ειρήνη και την ασφάλεια στην Αφρική. Όλα αυτά τα θετικά δεν θα πρέπει να κρύβουν τα αρνητικά στοιχεία όπως είδαμε στην πρόσφατη έκθεση Μόρ Ιμπραχήμ, έχουν χαθεί ευκαιρίες και η αύξηση του ΑΕΠ που μπορεί να υπάρχει δεν έγινε βιώσιμη οικονομική ευκαιρία για τον πληθυσμό και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ε, επίσης το δημογραφικό είναι ανησυχητικό. Η Αφρική επίσης ε, χυμάζεται από πολλά προβλήματα ασφαλείας και σε πολλές χώρες όχι μόνο οικονομικά. Για τη δημογραφία δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ξέρετε τις προοπτικές. Αναμένεται να διπλασιαστεί ο, ο, πληθυσμός μέχρι το 2050 από 1,2 δισεκατομμύρια σήμερα σε 2,4 δισεκατομμύρια. Ε, είναι μεγάλη ανησυχία αλλά και μεγάλη ευκαιρία αν τις αδράξουμε θα πρέπει οι νέοι να πιστεύουν ότι θα έχουν μέλλον στην Αφρική και αυτό δεν σημαίνει μόνο επιχειρήν και θέσεις εργασίας, αλλά να ζουν σε ειρήνη, ασφάλεια και σε ένα περιβάλλον που να μπορούν να αναπτυχθούν. Επίσης, οι επιχειρηματίες ε, ανησυχούν και δεν επενδύουν όταν είναι ανασφαλές το περιβάλλον. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν πώς συνδέεται η οικονομία με την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ως ενιαία αγορά παραμένει ο παριθμόν ένα επενδυτής αλλά και εμπορικός εταίρος στην Αφρική και πάροχος αναπτυξιακής βοήθειας. Το 2018 ήμασταν επίσης ε, ο πρώτος δωρητής της Αφρικανικής Ένωσης που καλύπταμε το μισό προϋπολογισμό της και με την διευκόλυνση 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε στείλει σε διάφορες ε, επιχειρήσεις όπως κυρίως αυτή στη Σομαλία. Εκτός λοιπόν από την δέσμευσή μας στην ειρήνη και την ασφάλεια με τη διευκόλυνση και τις δικές μας ε, αποστολές, στρατιωτικές και πολιτικές, ε, η εστίαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας, επενδύσεις, δεξιότητες, παιδεία, όπως ορίστηκαν πρόσφατα όλα αυτά στην αντίστοιχη διάσκεψη και ε, στην πρωτοβουλία την Ευρωπαϊκή για τις επενδύσεις. Θα ήθελα λίγο να σας μιλήσω και για την Κίνα και την παρουσία της στην Αφρική. Η Κίνα είναι σημαντικός παίκτη και οικονομικός και εμπορικός και ε, γενικότερα. Ε, τα τελευταία 20 χρόνια η Κίνα έχει γίνει πρωταγωνιστής ε, οικονομικός στην Αφρική. Σε κάποιες χώρες ε, έχει ξεπεράσει την, Αφρική, την Ευρώπη, συγγνώμη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ως επενδυτής και τέρος. Η Ρωσία, η Ινδία και ε, οι χώρες του Περσικού κόλπου επίσης είναι νέοι οικονομικοί παράγοντες και αναμένεται να επεκταθεί ακόμα η παρουσία της Κίνας στην Αφρική. Ωστόσο, δεν βλέπουμε με ποιο τρόπο, δεν βλέπουμε όλους αυτούς τους πρόσφατους ε, παράγοντες ως ανταγωνιστές μας. Μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην ασφάλεια της Αφρικανικής Υπήρου. Η Αφρική αυτό που χρειάζεται είναι να, καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες της και δεν μπορεί καμία χώρα να το κάνει αυτό. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή τους τράπεζα, για να φτάσουν στους στόχους της, τους βιώσιμους του ΟΗΕΤ μέχρι το 2030, χρειάζονται 130 δισεκατομμύρια ετησίως οι αφρικανικές χώρες. Τα κονδύλια αυτά ε, ε, έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των πόλεων και της υπαίθρου, πρόσβαση σε νερό και σε αποχέτευση, αλλά και συγκοινωνίες και μεταφορές. Ε, χρειάζονται για να αναπτυχθούν αυτές οι δομές ε, και τους παραδοσιακούς και τους νέους χρηματοδότες. Ε, νοσοκομεία, δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες, ε, χρειάζονται πολλά έργα υποδομής και άλλα. Άρα, στην Αιθιοπία, στην Κένια έχουν δημιουργήσει πολλά εργοστάσια οι Κινέζοι και πολλές θέσεις εργασίας. Εμείς έχουμε συμφέρον ε, οι ξένες εταιρείες να σέβονται τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς για τους διαγωνισμούς, ε, τις διεθνείς προδιαγραφές για την εργασία, τη διακυβέρνηση, την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να συνεισφέρουμε ε, στην ευημερία των αφρικανικών κρατών, αντί να επιδεινώσουμε τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Υπάρχει μια πλατφόρμα τώρα εκεί με την Αφρική για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε σχέδια κοινού συμφέροντος και ένα από αυτά είναι η Αφρική. Έχουμε αρχίσει ένα διάλογο με την Κίνα για να εμβαθύνουμε την αμοιβαία μας κατανόηση για την Αφρικανική Ήπειρο και να μπορούμε να την υποστηρίξουμε για την ασφάλεια και την ειρήνη και οικονομικά. Είναι κοινό το συμφέρον μας, ε, ώστε η Αφρική να είναι σταθερή, ευημερούσα ε, και ε, σε ειρηνική κατάσταση. Συνεργαζόμαστε και στα ναυτικά. Από το 2008 συμμετέχει η Κίνα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξασφάλισης της ναυσιπλοείας. Και κατά καιρού έχει συμμετάσχει στην επιχείρηση Αταλάντα, ε, συνοδεύοντας στρατιωτικά προς τη Σομαλία σκάφη που μετέφεραν παγκόσμια επιστηστική βοήθεια δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει χώρος για περισσότερη συνεργασία που πρέπει να διερευνήσουμε μαζί με την Κίνα από κοινού για να βοηθήσουμε τις χώρες της Αφρικής για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, για τη διακυβέρνηση ε, των ευρωπαϊκών και κινέζικων ιδιωτικών εταιριών στην Αφρική. Ως ΕΙΕΔ θέλουμε να συνεργαστούμε περισσότερο με την Κίνα για να εδραιώσουμε και να βελτιώσουμε τα επιτεύγματα ε, που έχουν ε, ήδη καταφέρει αλλά και τα επόμενα στα οποία προσδοκούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσουμε τη γενική συζήτηση, η οποία δυστυχώς θα είναι πολύ σύντομη, ο κύριος Γιολάινεν θα πάρει τον λόγο, που είναι πρόεδρος αντιπροσωπείας. Καλημέρα, πρόεδρε. Χαίρομαι που αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα Έχουμε, το έχουμε συζητήσει και στην αντιπροσωπεία για τη σχέση με την Κίνα δύο φορές και είχε έρθει ξανά ο κύριος Βγαλόγκα. πρώτα θα περάσω στα γερμανικά. Ε, λοιπόν, εμείς μπορούμε να λυπόμαστε που είναι τόσο δραστήρια η Κίνα στην Αφρική, αλλά να το αλλάξουμε δεν μπορούμε. Είναι γεγονός αυτό. Ε, χτες μόλις επέστρεψα από την Ιγυρία όπου δεν έγιναν τελικά εκλογές αλλά και στο Λάγος και στην Αμπότζα και παντού στην Αφρική βλέπουμε κινέζικες εταιρείε να κατασκευάζουν δρόμους και αυτοκινητοδρόμους. Οι Ευρωπαίοι είναι πόντες, αόρατοι. Οι υποδομές τώρα στην Αφρική κατά κύριο λόγο κατασκευάζονται από κινέζικες ε, εταιρείε. Και εδώ υπάρχει ένα ειδικό θέμα, το θέμα ε, των ε, συμφερόντων ασφαλείας των κινέζικων και των ευρωπαϊκών στην Αφρικανική Ήπειρο. Χαίρομαι που έχουμε αυτό το διάλογο για θέματα ασφαλείας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά πιστεύω ότι παρόλα αυτά υπάρχει δυναμικό. Γιατί όσο εντείνεται και αυξάνεται η παρουσία της Κίνας στην Αφρική, τόσο μεγαλύτερο συμφέρον έχουν να είναι ασφαλής ήπειρος. Εκεί υπάρχουν συνέργειες που μπορούμε να αναπτύξουμε και ε, συμπίπτουν τα συμφέροντά μας. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι σε σχέση με αυτά που είπατε. Και η Κίνα κάποια στιγμή θα ανακαλύψει ότι στην Αφρική ε, γίνονται πόλεμοι για το νερό, ε, για την κατανομή των γεών, για την αναδιανομή των γεών και το θέμα είναι πόσο μπορούμε εμείς να ε, φέρουμε στο πλευρό μας την Κίνα για τους στόχους της βιώσιμης, ε, βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ίσως όχι και για τους 17, αλλά ο κύριος Βιλαλόγκα μίλησε για το διάλογο σχετικά με το κλίμα. Υπάρχουν εκεί δυνατότητες. Επίσης, νομίζω ότι στο στενό στρατιωτικό τομέα θα πρέπει να αναζητήσουμε τομεί συνεργασίας με την Κίνα. Ε, γιατί συμμετέχουν στις αποστολές του ΟΗΕ, αλλά ε, ε, αποφεύγουν να μπουν σε περιοχές με ένοπλες σειράξεις. Στους κιανόκρανους πολλές φορές ε, η Κίνα αρνείται να συμμετάσχει. Δεν στέλνει τους δικούς στρατιώτες γιατί είναι πολύ επικίνδυνα. Λέει δεν πειράζει να στείλουμε κανέναν άλλον καλύτερα. Είπατε ότι η Κίνα ε, είναι ο δεύτερος εξαγωγές όπλων προς την Αφρική. Ε, και εκεί θα πρέπει να υπάρχει μεγάλος χώρος για συνεργασία. Πού καταλήγουν αυτά τα όπλα. Τα μεταπολούν γιατί μετά μπορεί αυτά να στραφούν ενδεχομένω και κατά των κινέζικων συμφερόντων. Υπάρχει ένα σύστημα διαφάνειας, κυκλοφορία των όπλων εκεί λογοδοσία υποχρεωτική. Και ένα τελευταίο, είπατε κύριε Βιλαλόγκα ότι προσπαθούμε και οι δύο να υποστηρίξουμε την Αφρικανική Ένωση και να την κάνουμε ακόμα πιο σταθερή και σε θέση να ορθοποδήσει στην ίδια της την Ήπεδρο και να φροντίζει για την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Εκείνα δεν είναι πάρα πολύ πρόθυμη εκεί. Εμεί είμαστε πάρα πολύ δραστηροί και μήπως να τη φέρουμε και αυτή σε αυτή την προσπάθεια θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Ευχαριστώ. Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις σας. Εγώ με άλλη ιδιότητα ασχολούμαι γενικά με την Αφρική αλλά καλό είναι και το συζητούμε εδώ στην υποεπιτροπή μας και έχουμε ε, αφιερώσει τη συζήτηση και σε αυτά τα θέματα ασφαλείας που θέλουμε να φωτίσουμε. Συμφωνώ ε, με το γιο Λάινεν και θέλω να συνεχίσω από κάποια στιγμή που ανέφερε Λέτε ότι είναι ο δεύτερος ε, εξαγωγέας όπλων η Κίνα στην Αφρική. Τι γίνεται με τον ελαφρύ οπλισμό ελαφρύς που σημαίνει ότι μεταφέρονται και εύκολα αυτά τα όπλα. Αυτός είναι ο υπαριθμόν έναν αποσταθεροποιητικός παράγων για πολλές περιοχές ε, που γνωρίζουν κρίση. Στο Σαχέλ, ας πούμε, ποιο είναι το ποσοστό κινέζικων όπλων που κυκλοφορούν ή στον Μπόκο Χαράμ ή ή σε άλλα χέρια. Ή μήπως είναι ρωσικά όπλα, αμερικανικά ή ευρωπαϊκά. Θα με ενδιέφερε να το γνωρίζω αυτό. Σε περίπτωση που είναι μεγάλο το ποσοστό των κινέζικων όπλων, αυτό θα μπορούσε να είναι αφορμή και για συζήτηση με την Κίνα. Ιδιαίτερα όταν δεν πέφτουν αυτά τα όπλα σε χέρια αναγνωρισμένων κυβερνήσεων, αλλά άλλων ε, μαχητών. Άλλη ερώτηση. Έχουμε εικόνα, αν κοιτάξουμε το χάρτη της Αφρικής, έχουμε εικόνα για το που προσπαθεί να αποκτήσει ναυτικές βάσεις η Κίνα, στοχευμένα οι αεροπορικές βάσεις, επιλέγει χώρες για να εγκατασταθεί. Υπάρχουν χώρες με τις οποίες έχουν επίσημες συμφωνίες αμυντικές ή ασφαλείας και θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι θα ανοίξουν και βάση κάποια στιγμή. Κάτι άλλο που θα με ενδιέφερε ιδιαίτερα ε, σχετικά με το ουράνιο. Ξέρουμε τι κάνει η Κίνα για το ουράνιο. Δραστηριοποιείται ιδιαίτερα γιατί γνωρίζω από την Αμίμπια ότι υπάρχουν κινέζικες εταιρείες που ασχολούνται με το ουράνιο και ιδιαίτερα σε αυτή τη χώρα που είναι μικρή και αεροκατοικημένη, δύο εκατομμύρια κατοίκους περίπου έχει η Ναμίμπια, υποτίθεται ότι είναι πάνω από 100.000 οι Κινέζοι. Αυτό δεν το έχω διασταυρώσει. Δεν φαίνονται στη χώρα, αλλά κάπου βρίσκονται αυτοί. Αν δείτε την πρεσβεία, είναι τεράστια. <laughs> Τελείως δυσανάλογη με το μέγεθος της χώρας. προφανώς θέλουν να ασκήσουν επιρροή. Υπάρχουν και άλλες ε, τέτοιες χώρες όπου είναι δυσανάλογα μεγάλη η παρουσία της Κίνας και σε ευαίσθητες περιοχές που έχουν και ευαίσθητες πρωτοσύλλες όπως είναι το ουράνιο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Άννα Γκόμες. Παρακαλώ, συνάδελφοι, σύντομοι να είστε. Συνολικά έχουμε ένα τέταρτο για αυτή τη συζήτηση. Μετά πρέπει να κλείσουμε αυτό το σημείο. Το 2008 ε, συνέταξα μία έκθεση στο Κοινοβούλιο, στα πλαίσια της Επιτροπής Ανάπτυξης, για την προοπτική της Ευρώπης και το ρόλο της Κίνας στην Αφρική. Και έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, και η Αφρική θα πρέπει να κάνουν μια τριγωνική σχέση. Όχι στην πλάτη των Αφρικανών, μαζί με τους Αφρικανούς, ούτως ώστε οι Αφρικανοί να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, να υπάρχει οικοδομή δυναμικού, και να υλοποιηθούν οι στόχοι, έλεγα τότε, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εμείς δεν ε, δεν είναι ότι δεν βλέπαμε ότι αυτό θα συνέβαινε, είναι ότι δεν θέλαμε να ασχοληθούμε και ότι έχουμε απεμπλακεί υπό από πολλές απόψεις από την Αφρική. Ε, θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις της ερωτήσεις που τέθηκαν, ειδικά για την πώληση όπλων. Είναι πραγματικά ε, όπλα μαζικής καταστροφής. Ε, μιλάμε για τα μικρά όπλα και ελαφρά όπλα. Η Κίνα είναι ο δεύτερος προμηθευτής. Όταν ε, εκδόθηκε η έκθεσή μου, ήταν ατυχή στιγμή γιατί ένα πλοίο τότε με όπλα για την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε είχε μπλοκαριστεί από την ε, ε, Ένωση στην Νότιο Αφρική και δεν ήθελαν να πάνε τότε στην Ζιμπάμπουε για να... γιατί θα υπήρχε πρόβλημα με το καθεστώ του Μουγκάμπε. Ναι, τα συνδικάτα μάλλον την το είχαν μπλοκάρει αυτό το πλοίο. Σήμερα έφτασα από την Αθιοπία, μόλις σήμερα το πρωί, όπου οι κινέζικες επενδύσεις είναι πάρα πολλές ε, και μακρές, ε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πόροι βέβαια. Αλλά αυτό συνδέεται και με την ε, ιδεολογική στήριξη του καθεστώτος που είναι καταπιεστικό. Αυτό το κάναμε και εμείς, υποστηρίξαμε αυτό το καταπιεστικό καθεστώς και τώρα υπάρχει αντίδραση βέβαια. Στην Αιθιοπία υπάρχουν φοβερές ε, βελτιώσεις ε, στο βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Υπάρχει στην Αντίσα Μπέμπα ένα τρένο που κυκλοφορεί, ε, είναι υπέργειο τρένο αυτό, το χτίσανε οι Κινέζοι. Έχει μια κυκλική πορεία. αν οι Ευρωπαίοι είχαν επενδύσει στην Αφρική, θα μπορούσαν να κάνει το ίδιο. Αλλά τώρα βλέπουμε τις αντιδράσεις αυτής της κατάστασης, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφθορά. Όλες αυτές οι διαφθορές, ε, σε αυτές τις διαφθορές γύρω-γύρω υπάρχει διαφθορά και ο κόσμος αντιδρά. Ο κόσμος έχει ε, βαρεθεί με την κατάσταση αυτή, με τη διαφθορά. Στηρίξαμε αυτό το ολοκληρωτικό καθεστώς, γιατί υποτίθεται θέλαμε να σταματήσουμε, ας πούμε, την κατάρρευση του καθεστώτο και άρα τη διάλυση τη Αφρική κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το καθεστώ οδηγούσε σε διαφθορά και αυτό το είδαμε σε πολλέ άλλε χώρε τη Αφρική. Το 2008 τότε αμφιβάλλανε αν οι Κινέζοι θα μπορούσαν να ασχοληθούν ε, στην Μοζαμβίκη και στην Αγκόλα, ας πούμε, ε, αλλάζει ο, ο κόσμος, αλλάζει η κατάσταση. Ε, οι Κινέζοι, ας πούμε, ε, ανακατεύονται με τον τόπιο πληθυσμό. Επίσης πρέπει να δούμε και την ε, στάση ε, με την, και τη διάθεση με την οποία γίνονται αυτές οι επενδύσεις ε, στην Αφρική και τη διαφθορά που προκαλούν και τις αντιδράσεις κατά συνέπεια. Θα σταματήσω όμως εδώ για να δώσω το λόγο στους ε, καλεσμένους μας. Θα ήθελα και εγώ να υποβάλω, λέει η Πρόεδρος, λίγες ερωτήσεις και στους δύο μιλητές. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για την ασφάλεια, για τη βάση του Τζιμπουτή. Υπάρχει μια διαφορά, παραδείγματο χάρη, οι Κινέζοι υποστηρίζουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας, έτσι, στην Αφρική και στην, στα αφρικανικά ύδατα και μας βοηθούν να καταπολεμήσουμε την ε, πειρατεία σε ειδικέ αποστολέ, Υπάρχει ένας ειδικό μηχανισμός, η Αταλάντα, η επιχείρηση αυτή. Από τη μία υπάρχει αυτό και από την άλλη υπάρχει απαγόρευση της ναυσιπλοείας στην Κινέζικη θάλασσα. Δεν υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Και στα στενά, ανάμεσα στην υπηρετική Κίνα και στην Ταϊβάν. Στα στενά της Ταϊβάν δηλαδή. Μία ερώτηση τώρα για τα μοντέλα που χρησιμοποιούν για να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή. Τι σχέση έχει η ασφάλεια με την κλιματική αλλαγή στην Αφρική. Και τι πολιτική χρησιμοποιεί η Κίνα στη δική της επικράτεια για να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή, στο δικό της έδαφος. Θα ήθελα να μου απαντήσετε με την ίδια σειρά η κυρία Βαλιαγνική πρώτα. Δεν Πολύ σύντομα, ε, γιατί ήμουν πολύ μακροσκελή στην πρώτη μου παρουσίαση, αλλά είχα πολλά να πω. Για τα μικρά όπλα, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Είναι τεράστιο θέμα, γιατί προκαλούν και καταπίεση, αλλά αυτά τα μικρά όπλα, όπως είπατε, μπορούν να πέσουν στα χέρια ομάδων και αυτό είναι παράγοντας αστάθειας, αύξηση της αστάθειας, ε, πρόκλησης προβλημάτων ε, σε επίπεδο ασφάλειας και για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. θα μπορούσαμε, αν γίνεται, εμείς να ενθαρρύνουμε την Κίνα να δεχτεί επιτέλους την ε, σύμβαση για τα συμβατικά όπλα. Το 2013 υπογράφτηκε, η Κίνα πήχε. Αυτά για τα μικρά όπλα. Για το Τζιμπουτί, η Κίνα δεν είναι η μόνη που έχει μια επιμελητιακή βάση στο Τζιμπουτί. Είναι τεράστια αυτή η αλλαγή στην ε, Κίνα, γιατί Μέχρι στιγμής αρνούνταν την ιδέα της στρατιωτική βάσης οι Κινέζοι. Το Τζιμπουτί ξέρετε πολύ καλά ότι έχει υπογράψει διάφορες συμφωνίες αναπτυξιακές κτλ. Ε, προσπαθεί να υποστηριχθεί από πολλές χώρες, όχι μόνο από την Κίνα, και γι' αυτό πολλές χώρες έχουν βάση στο Τζιμπουτί. Αλλά η επιμελητιακή βάση της Κίνας στο Τζιμπουτί είναι τεράστια και θα μπορούσε να δεχτεί τεράστιο προσωπικό και αυτό συνδέεται με τα άμεσα συμφέροντά τους ε, σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό που έχουν και την ανάγκη να κενώσουν τον πληθυσμό ή την πρόσβαση στους πόρους. Η Κίνα θέλει να χτίσει στην Ιγερία μία άλλη βάση, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Έχουν ξεκινήσει στρατιωτικές ασκήσεις με την Ιγυρία ε, γίνεται τεράστιος εταίρος η Κίνα της Νιγηρίας λόγω των, της ενέργειας, των πόρων που έχει και η Κίνα πραγματικά είναι πολύ παρούσα σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα ερώτημα. Η Κίνα συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο την ανάγκη να ελέγξει περιβαλλοντικά προβλήματα και συνειδητοποιεί το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, ακόμα και στο εσωτερικό της Κίνας. Το μεγάλο πρόβλημα όμως που έχουμε με την Κίνα είναι ότι από τη μία γίνονται μεγάλες δηλώσεις, αλλά από την άλλη το σύστημα μια και δεν υπάρχει ελεύθερος τύπος, δεν υπάρχει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, δεν υπάρχουν οι βάσεις ουσιαστικά για να βελτιωθεί η κατάσταση. Έχουμε απλώς ηχηρές δηλώσεις. Και αν η εξουσία θέλει να κάνει κάτι η ηγεσία θέλει να κάνει κάτι για το, την κλιματική αλλαγή, θα το κάνει. Αλλά δεν υπάρχει κανένα έλεγχο. Και η ίδια λογική, η ίδια κουλτούρα εξάγεται παντού, οπουδήποτε είναι παρούσα και δραστηριοποιείται η Κίνα. Και στην Αφρική προφανώ. Ε, και στη Λατινική Αμερική βεβαίω. Που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα λόγω των σχέσεών τη με την Κίνα. Μην ξεχνάτε τι γίνεται στην Βενεζουέλα σήμερα. Η Βενεζουέλα ήταν βασικό εταίρο τη ε, Κίνας η στήριξη της Κίνας, μιας χώρας από την Κίνα, δημιουργεί, σε, προβλήματα. Όταν μιλάμε για το αναπτυξιακό μοντέλο της Κίνας, το μοντέλο που μας παρουσιάσει, μην ξεχνάμε την πραγματικότητα αυτού του μοντέλου. Και η πραγματικότητα ποια είναι, συνοψίζεται στην πραγματικότητα της Βενεζουέλας γιατί έχουν απαντηθεί πολλά ερωτήματα και εγώ θα απαντήσω τα υπόλοιπα. Ο κύριος Λάινεν. Ρωτήσατε ή αναφέρατε μάλλον κάτι με το οποίο συμφωνώ. Όσο περισσότερο επενδύει η Κίνα και δραστηριοποιείται στην Αφρική, τόσο περισσότερο συμφωνούμε και για άλλα θέματα, και για την ειρήνη και για την ασφάλεια και ανησυχούμε για την παρουσία της ε, εκεί, αλλά το βλέπουμε και ως ευκαιρία για να συνεργαστούμε σε κάποια θέματα οικονομικής διακυβέρνησης, χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης, γιατί ε, και αυτό επηρεάζει τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις. Ε, και σε σχέση με τα όσα ρώτησε η κυρία Γκόμενς για την τριγωνική συνεργασία, μακάρι να είχαμε ε, θέλουμε πολύ περισσότερο να συμμετέχουν για την ειρήνη και την ασφάλεια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Αφρικανοί δεν έχουν ενθουσιαστεί ε, ε, από το ενδεχόμενο να συνεργαστούμε εμείς με την Κίνα. Και τον κύριο Κάλερ βλέπω πολλές φορές στις συνεδριάσεις ΣΑΚΕ ε, κάθε φορά που προσπαθήσαμε να αφαιρθούμε στην Κίνα ε, δεν ε, ακούσαμε μια θερμή ενθουσιώδη αντίδραση, μάλλον το αντίθετο από τις αφρικανικές χώρες. Εκείνοι θέλουν να συνεργάζονται με την Κίνα και με εμά ξεχωριστά. Δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε και ελπίζω να υπάρξει κάποια πρόοδος. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δεν έχουμε προβλέψει δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Είναι πολλά τα θέματα ακόμα στη μέση διάταξη και έχουμε κάποια χρονική πίεση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και τους δύο διακεκριμένους ομιλητές μας, αλλά ε, και τα μέλη που πήραν το λόγο. για να κλείσω αυτό το σημείο. Παρακαλώ. Ας χειροκροτήσουμε όλοι μαζί τους ομιλητές μας. Thank you. We start immediately. Λοιπόν, συνεχίζουμε αμέσως με το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, που είναι ε, θέματα ασφαλείας, πτυχές σχετικές με την ασφάλεια στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασίας.